χρόνο και μεταξύ εσωτερικών και εσωτερικών ανισοτήτων. Ευχαριστούμε. Να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία από τον ΕΟΧ, του συναδέλφους από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία, που είναι καθώς και παρατηρητές από την ε, ε, Ελβετική Συνέλευση που βρίσκονται στην αίθουσα. Από την ΕΖΕΣ λοιπόν όλοι οι παρατηρητές που θα συμμετάσχουν στην ε, συνάντηση σήμερα και αύριο ελπίζουν, ελπίζω ότι θα μπορέσουν ε, να δώσουν αποτελεσματικό έργο με τη συνεισφορά τους και να βοηθήσουν στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας καθώς και την ε, καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Now I give the floor to our next speaker. Επόμενος Ομιλητής η κυρία Φαν Μπρέμπτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντας κανείς τη σημερινή συζήτηση διαπιστώνει το εξής. Ε, όλες οι πολιτικές ομάδες σχεδόν ζητούν οικονομική διακυβέρνηση. Είναι φαινομενική αυτή η ομοφωνία γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο